ασφάλειά μας είναι η αχανή λύνωτη μαζική μετανάστευση, η Ισλαμιοποίηση, οι Ισλαμικές επιθέσεις που απορρέουν από τη μαζική μετανάστευση. Και τώρα η ΕΚΕΠΑ και η ΕΠΑ δεν έχει αντιμετωπίσει ούτε έχει μειώσει την απειλή αυτή. Το αντίθετο παρακαλώ να μην θίξετε την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών και να μην αναγκάσετε σε συνεργασία τα κράτη-μέλη. βεβαίω για το υλικό, το στρατιωτικό και και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών όλα είναι καλά και αποτελεσματικά στην καταπολέμηση τη μεγάλη, όπω είπα απειλή, που είναι η μαζική μετανάστευση, ο εξισλαμισμό και η τρομοκρατία. Οι συστάσει μας λοιπόν είναι σαφεί. Σταματήστε τη διεύρυνση της Ένωσης, σταματήστε την προσέγγιση με την Τουρκία και συνεργαστείτε με εταίρου όπως είναι η Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Ο λόγος του κύριο Βέιμερς ε, από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, όταν ήρθα πριν από πέντε χρόνια στις Βρυξέλλες, είχα μια σαφή εικόνα για το τι εστίκει είναι εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Ε, εγώ φανταζόμουν την διακυβερνητική συνεργασία, διακρατική συνεργασία για κοινέ επιχειρήσεις. Αλλά ε, η ε, Σουηδία και άλλες χώρες να μπορούν να έχουν την ανεξάρτητη διεθνή τους εξωτερική πολιτική. Γρήγορα όμως ανακάλυψα ότι πολλοί αντιτίθενται ε, στεναρά σε αυτή την ε, ιδέα. Ήθελαν περισσότερη στρατιωτική ε, δύναμη και ισχύ με φεντεραλιστικές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν και αντιαμερικανικές δυνάμεις. Να έρθουν περισσότεροι τομείς πολιτικής, να εκχωρηθούν περισσότερες εξουσίες στις Βρυξέλλες, όπως και αλλού. Έχουμε διαβάσει για στρατιωτικοποίηση, για όπλα, τώρα για αποφάσεις όχι με ομοφωνία αλλά με ενισχυμένη πλειοψηφία. Δεν υπάρχει αρκετή υποστήριξη για αυτή την πρόταση. Από τους μη εγγεγραμμένους τώρα, Τζέικ Πού. Όχι, αποσιάζει ο κύριος Μιλιάν Μον. Ε, ο λόγος σας για ένα λεπτό. Ο προηγούμενος ομιλητής είναι απόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολιτικό όραμα που βασίζεται στο κράτος δικαίου και στην επικράτηση του δικαίου. Ιδρύθηκε για να ξεπεραστούν οι ακραίοι εθνικισμοί. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει χώρος για αυτούς που δεν σέβονται το νόμο και το κράτος δικαίου <clears throat> ε, που ε, μάλιστα ε, διαφεύγουν κιόλας ε, του νόμου. Εδώ έχουμε έναν φυγά από την δικαιοσύνη του οποίου η μοίρα είναι τα ίδια τα δικαστήρια που θα δώσει λογαριασμό. Τώρα, περνάω στην συζήτησή μας. Ο κόσμος είναι πολύ περίπλοκος και ε, πολυπολικός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πέσει στην παγκόσμια σκακέρα για να προασπίζει τις αξίες της και τα ε, συμφέροντά της. Θα πρέπει να είναι ένας παίκτη αξιόπιστος. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μακάλιστερ και τον κύριο Ντόνζο για τις εκθέσεις τους, που είναι πλήρης ιδιαίτερα σε αυτή του κυρίου Ντανζό αναφέρεται πολύ και η διάσταση της άμυνας που είναι όλο και πιο σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ευτυχώ έχουμε κάνει πρόοδο. Ευχαριστώ. Ο κ. Μίξερ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε και εξακολουθεί να είναι ένα σχέδιο ειρήνης σε θέματα άμυνα έχουν καθυστερήσει λίγο. Γι' αυτό το λόγο εξακολουθούν να υπάρχουν συνάδελφοι ε, που δεν αισθάνονται άνετα με το να συζητάμε θέματα άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν να τα αναφέρουμε στην ίδια φράση. Υπάρχουν δύο ειδών επικριτές. Πρώτον, αυτοί που φαίνεται ότι πιστεύουν ειλικρινά πως ε, όλες οι συγκρούσεις στον κόσμο μπορούν να επιληθούν χωρίς τη χρήση βίας και όπλων. Και οι δεύτερη κατηγορία που λέει ότι θα πρέπει ε, όλες οι, όλες συγκρούσεις να ε, αφαιθούν στα χέρια των ΗΠΑ και των άλλων μεγάλων δυνάμεων. Ε, Δυστυχώ δεν συμφωνώ ούτε με την πρώτη με τη δεύτερη. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε όλε τι συγκρούσει να τι λύσουμε με ειρηνικά μέσα. Δυστυχώ. Ε, πολλοί από εμά θεωρούν ότι είναι πολύ κακό που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κόσμο, παρόλο ότι έχουμε μια πολύ φιλόδοξη παγκόσμια στρατηγική. Για να μπορούμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο, πρέπει να έχουμε στρατιωτικέ ικανότητε που δεν είναι και ούτε δωρεάν ούτε φθηνέ. Αν λοιπόν <clears throat> θέλουμε να παίξουμε ένα πιο σοβαρό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να αφιερώσουμε και τις κατάλληλες ε, ε, υποδομές. Ευχαριστώ κύριο Σαουστρεβίτσιους από την ομάδα Renew. Είπατε εκπρόσωποι, συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές για την εξαιρετική τους εργασία σήμερα. Η ΚΕΠΑ και, και η πολιτική ασφάλεια και άμυνας θα πρέπει να συνοδεύονται από αλλοκατανόηση των ε, προκλήσεων και από κοινή δράση. Θα πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων μας και των αμυντικών για να είμαστε σε θέση ε, να αντιμετωπίζουμε στην άμεση γειτονία μας τις κρίσεις που προκύπτουν. Οι πολιτικές γειτονίας προς Ανατολά και προς Νότο θα πρέπει να συνδυάζουν πολιτική, οικονομική άμυνα, ε, ασφάλεια αλλά και άμυνα ταυτόχρονα. Έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε σε συνεργασίες με ε, τους δημοκρατικούς εταίρους και γειτονές μας. Δυστυχώς ο κατάλογος αυτών των δημοκρατικών κρατών όλο και συρρυκνώνεται. Επιπλέον, το οικονομικό συμφέρον δεν θα πρέπει να επισκιάζει ε, τα θέματα ασφαλείας. Είναι πραγματικά λυπηρό και απογοητευτικό να βλέπουμε έργα τύπου Nord Stream 2 ε, και να κυριαρχούν τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά η Ρωσία έχει ε, γεωπολιτικές βλέψεις και καταστροφικές σε Λιβύη και Συρία. Η κυρία Ζόφκο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η νέα Κομισιόν θέλει να είναι γεωπολιτική. Ε, ε, σε παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι ε, καταπληκτική ευκαιρία αυτές οι δύο εκθέσεις για να δούμε και να διατρανώσουμε και πάλι τη θέση του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να συγχαρώ τους κυρίους Μακάλιστερ και Ντανζάν. Είναι εξαιρετικές οι εκθέσεις τους και στις δύο εκθέσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαφώς αναγνωρίζει και υπογραμμίζει ρητά ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που να μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Για μένα κομβικό εδώ είναι οι σχέσεις ε, της Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Εκτός από το γενικό στόχο ε, τη ΚΕΠΑ θα πρέπει να καθοδηγήσουμε τις χώρες αυτές προς την ένταξη που τους αξίζει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ε, ε, Διάφορε αποστολές όπως είναι η Αλθέα στη Βοσνία Ζεγοβίνη και είναι η πρώτη ευρωπαϊκή που δουλεύει καλά και παίζει ε, κομβικό ρόλο για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ένωσης και της Υπήρου μας. Εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δείξουμε στήριξη για την ευρωπαϊκή προοπτική της περιφέρειας των Βαλκανίων. Και με διάφορα προενταξιακά μέσα. Ω εισηγήτρια για το μεσο η ΙΠΑ3 ε, πρέπει να τονίσω ότι θα πρέπει να ελέγχουμε και να καθοδηγούμε το πρόγραμμα αυτό. Στην άμεση γειτονία μας, στα Δυτικά Βαλκάνια, έχουμε χώρες που ανήκουν στην Ευρώπη και είναι σημαντικό το θέμα ασφαλείας. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια που ξεκινήσαμε για τη διεύρυνση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σούστερ, ο οποίο ε, μπορεί να μιλήσει και λίγο παραπάνω. Θα μιλήσει εκ μέρου των σοσιαλδημοκρατών. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι επιθυμούμε εμβάθυνση της πολιτικής ασφάλειας. Υπό τον Τραμπ οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν γίνει ένας απρόβλεπτος τέρος. Η Ρωσία θεωρεί ότι η στρατιωτική επέμβαση είναι κάτι φυσιολογικό για να προστατεύει τα συμφέροντά της και πάρα πολλές διενέξεις ε, καταλήγουν σε ε, πόλεμες συγκρούσεις. Αλλά στην Ευρώπη όχι μόνο πρέπει να συνεργαστούμε πιο ε, στενά, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εδώ υπάρχουν κάποιε διαφορέ. Δεν καταλαβαίνω γιατί η εντετικοποίηση τη συνεργασία ε, πρέπει να συνοδεύεται με ουσιαστική και ριζική αύξηση των ε, αμυντικών προπολογισμών. Οι στρατιωτικέ δαπάνε των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνουν πολύ περισσότερε από αυτέ της Ρωσία. Δεύτερον, οποτεδήποτε θέλουμε να έχουμε του εξοπλισμού αποτελεσματικότερου, χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα από ό,τι σήμερα για τους εξοπλισμούς. Και τρίτον, οι συγκρούσεις ε, κατά κανόνα ε, διεξάγονται και δεν μπορούν να επιληθούν ούτε με στρατιωτική επέμβαση, ούτε με εξοπλισμού. Χρειαζόμαστε μια πολιτική που να βασίζεται περισσότερο στη διπλωματία, στην ενίσχυση των αφοπλισμών και χρειαζόμαστε και περιορισμό των ε, εξοπλισμών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρίως ε, Κιούτσουκ ε, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Μπορέλ, Ευχαριστώ τους συγητές για την έκθεσή τους. Η πολυμερή ε, τάξη αλλάζει. Ε, πλέον έχουμε υβριδικούς πολέμους, τρομοκρατία. Αυτή λοιπόν η περίπλοκη κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ίσως να μην μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες, αλλά ούτε και το κράτος δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την διεθνή συνεργασία. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, η Αφρική και οι γείτονές μας. Όλοι αυτοί χρειάζονται την υποστήριξή μα γιατί τα γεγονότα που διαδραματίζονται εκεί έχουν άμεση επιπτώσει εδώ. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική τη τη γειτονία, στηρίζοντας ε, την εδαφική ακαιρεότητα, τη σταθερότητα, τη συνεργασία με όλε τι προαναφερθήσει χώρε. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αξιόπιση στρατηγική στα Δυτικά Βαλκάνια. Η διεύρυνση θα συνεχίσει να είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία μα τη εξωτερική πολιτική. Πρέπει να τα καταφέρουμε σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί και να διατηρήσουμε ανοιχτή την προοπτική των ε, Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κιούμπιλους για ένα λεπτό εκ μέρους του ΕΛΚ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις εξαιρετικές εκθέσεις τους. Δεύτερον, έχω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, πρώτη παρατηρήση, πρώτο στόχο τη πολιτικής, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σαφή. Η Ευρώπη πρέπει να ζήσει ειρηνικά και να δημιουργήσει επιτυχίες και στις γειτονικές χώρες όπως για παράδειγμα στην Ουκρανία. Δεύτερον, είναι καιρός να περάσουμε στην ε, ενισχυμένη πλειοψηφία. Γιατί ε, με την ε, ομοφωνία καταλήγουμε απλώς να κάνουμε κενές δηλώσεις. Τρίτον, όταν μιλούμε για την ευρωπαϊκή ε, στρατηγική αυτονομία τη ε, Ευρώπη εντό του ΝΑΤΟ, πρέπει να είμαστε πιο σαφεί. Χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ και την αμερικανική ε, πυρηνική ισχύ στην Ευρώπη αποτρεπτικά εναντί της Ρωσίας. Όμως θα πρέπει να έχουμε ισχυρή στρατιωτική και διπλωματική δύναμη για να ισχυροποιήσουμε και να σταθεροποιήσουμε τη γειτονιά μας. Merci. Ο κύριος Γκλουξμάν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές. Η μύθη της δεκαετίας του 90 για το τέλος της ιστορίας ή για την ευτυχή παγκοσμιοποίηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών ανήκουν στα σκουπίδια της ιστορίας. Σήμερα θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θα παραμείνουμε αιώνιοι έφηβοι με λόγια μόνο και σε κάθε κρίση ε, τρέχουμε στην αγκαλιά του μπαμπά, ε, του Αμερικάνου. Ή αν θα ενελικιωθούμε. Αν θέλουμε να ενελικιωθούμε και να χτίσουμε την ε, στρατηγική ανεξαρτησία της Ευρώπης και να έχουμε και βάρος σε αυτόν τον επικίνδυνο κόσμο, θα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να ε, οικοδομήσουμε αυτή την ευρωπαϊκή άμυνα. Είναι αφόρητη η κατάσταση. Δεν μπορούμε να έχουμε στο Σαχέλ Γάλλους στρατιώτες που να σκοτώνονται ε, χώρες που να δίνουν πολλά χρήματα από τον προπολογισμό για να χτίσουν την ευρωπαϊκή άμυνα και κάποιες όλες ε, χώρες θεωρούν ότι το τέλος της ιστορίας είναι ένας μύθος που ισχύει. Και ευχαριστώ του συγητέ για τα σταράτα λόγια τους. Ευχαριστώ πολύ. Λούκα Μάντελ τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Εγώ θα υπερψηφίσω και τις δύο εκθέσεις και ευχαριστώ τον ε, Μακάλιστερ και τον Τανζάν για τις εκθέσεις αυτές, ιδιαίτερα για τη διατύπωση που αφορά την κατάσταση ασφαλείας γύρω από την Ευρώπη, ότι έχει επιδεινωθεί δραματικά. Δηλαδή αυτό σημαίνει για μας καθήκον και αποστολή και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλος ιδιαίτερος για το Συμβούλιο. Και για αυτό το λόγο και για άλλου χρειαζόμαστε μια νέα συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, είναι απαρχιωμένη πλέον η συνθήκη τη Λισαβόνα. δεν αντέχει στι σημερινέ προκλήσει. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να είναι πιο ισχυρή προ τα έξω και πιο ελεύθερη προ τα μέσα. Ναι, νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη λοιπόν θα πρέπει να προβλέπει την κατάργηση τη ομοφωνία σε θέματα εξωτερική πολιτική στο Συμβούλιο ε, και σε θέματα ασφαλεία. Επιτέλου να μπορεί η Ευρώπη να παίρνει αποφάσει. Και όπω συμβαίνει και στη ζωή του καθενός προσωπικά, το να μην παίρνει απόφαση είναι η χειρότερη απόφαση που μπορεί να πάρεις. Αναμένω λοιπόν και νομίζω ότι μιλώ εξ ονόματο πολλών βουλευτών να ασχοληθούμε ιδιαίτερα για αυτή την πολιτική. Ε, η Επίτροπη, όπως προβλέπετε, από την επιστολή αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, παρακαλώ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Στάθειας πολλαπλασιάζονται γύρω μας αυτή η νέα πραγματικότητα αναδεικνύει την ανάγκη για ενιαία εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα και ασφάλεια. Δυστυχώ είμαστε μακριά από αυτόν τον στόχο με ευθύνη ισχυρών κρατών και αυτό έχει πολύ σοβαρέ συνέπειε σήμερα. έχετε επιτρέψει με την αβουλία σα θέματα υψή τη σημασία για την ασφάλεια των λαών τη Ευρώπη να τα χειρίζονται ο τραμπ ο πούτιν και ο ερντογάν. κάποιοι παραγνωρίζετε αυτή την οπτική γιατί απλά δεν συνορεύεται με χώρε που δεν σέβονται το διεθνέ δίκαιο. η ελλάδα παραδείγματο χάρη ξοδεύει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προπολογισμού τη για εξοπλισμού μειώνοντα τη χρηματοδότηση για το κοινωνικό κράτο την υγεία και την παιδεία. δεν μπορεί όμω να υπομίζονται κάποιοι μόνοι του όλο το βάρο προστασία των κοινών συνόρων απέναντι σε κοινέ απειλέ. ήρθε η ώρα να κάνετε όσα δεν κάνατε στο παρελθόν. είναι θέμα δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. η ένωση να γίνει στρατηγικά αυτόνομη και να αναπτύξει τις δικές της αμυντικές δομές κάτι που σήμερα φαίνεται ουτοπία είναι μονόδρομος για το μέλλον. Ο κύριος Κρίς Πέτερς, ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Μπορέλα, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να συγχαρώ τους δύο συζητητές για την εξαιρετική τους έκθεση και βεβαίως ε, ε, υπάρχουν ε, παγκοσμίω μεγάλες αναταράξεις, η παγκόσμια τάξη κλονίζεται, οργανώσεις όπως το ΝΑΤΟ δεν αποτελούν πλέον πυλώνα σταθερότητας, οι συμφωνίες ε, καταγγέλλονται, παραβιάζονται κτλ. Χρειάζεται μια πολυμερή συνεργασία. Αυτή είναι η καλύτερη διεθνής και παγκόσμια τάξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει γρήγορα να γίνει αυτόνομη στρατιωτικά. Έχουν γίνει βήματα επιτάχυνσης. Για να έχουμε αυτή τη στρατηγική αυτονομία όμως στην άμυνα, χρειάζονται προσπάθειες. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Καλό τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν έτσι ώστε στο τέλος της παρούσης θητείας να έχουμε μια αποτελεσματική λειτουργική επιχειρησιακή ευρωπαϊκή άμυνα στις 8 Μαΐου μάλλον 26 Μαΐου του 2019 ψήφισαν οι Ευρωπαίοι πολίτες προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όλεκας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι οι συγητέ έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πραγματικά να παίζει σημαντικό ρόλο στο σημερινό κόσμο με τι απειλέ, εάν έχουμε τη φιλοδοξία να μην είμαστε διακοσμητικοί σε αυτόν τον κόσμο, θα πρέπει να ενισχύσουμε τι οικονομικέ και διπλωματικέ μα δραστηριότητε, να αποφύγουμε κλιμάκωση σχετικά με το θέμα των συνόρων. Αλλά δεν αρκεί αυτό, γιατί στη γειτονιά γειτονιά μας έχουμε απρόβλεπτα καθεστώτα Συρία, Ιράκ, Ιράν και Ρωσία. Πρέπει να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας, ε, την αντοχή μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα αυτοκρατικά καθεστώτα ε, κατανοούν το παιχνίδι μόνο με ισχυρούς ε, παίκτες και αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά ισχυροί παίκτε, πρέπει να εκταμιεύσουμε πόρους για να έχουμε ικανοποιητικέ υποδομές. Και το 2% ε, του ΑΕΠ σε κάθε χώρα. Θα πρέπει να ισχύει αυτό. Αυτός είναι ο στόχος. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κύριο Πόξκο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τους εισηγητέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουγγαρία στηρίζουν την ακαιρεότητα και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ε, τι διαπραγματεύσεις για να επανέλθει σύντομα ειρήνη σε αυτή τη χώρα το ε, καθεστώς της Νορμανδίας. Ε, αυτή η πλατφόρμα βοήθησε στο να έχουμε ανταλλαγή φυλακισμένων. Ε, υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλές εντάσεις. Η προηγούμενη κυβέρνηση ακολούθησε μια εθνικιστική πολιτική και τα δικαιώματα των μειονοτήτων περιορίστηκαν ο νυν πρόεδρος ε, πλέον ε, καλεί τους πολίτες της Ουκρανίας ε, να συνεργάζονται και αυτό είναι μια θετική, ένα θετικό μήνυμα. Ελπίζω ότι αυτό θα φέρτε και στο σύνταγμα της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη ειρήνης στις γειτονικές, στις γειτονικές περιοχές, αλλά πρέπει να τηρούνται και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ο κ. Μπίλτσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για τις εξαιρετικά ισορροπημένες εκθέσεις τους. Ε, να κάνω μερικέ ε, ε παρατηρήσει για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική, ασφάλειας. Ε, χρειάζεται να προσπίσουμε τα ευρωπαϊκά στρατηγικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο και θα πρέπει ε, ιδιαίτερα να στηρίξουμε τη γειτονία μας. Η γειτονία μας, η γειτονιά μας είναι το σημείο στο οποίο θα κριθεί η πολιτική αυτή. Ε, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Τουρκία, ούτε η Κίνα ε, δεν πρέπει να πετύχουν στα Δυτικά Βαλκάνια πριν από εμά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει παίξει ρόλο, αλλά από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Κομισιόν και με τα κράτη-μέλη προκειμένου να πετύχουμε απτά αποτελέσματα επιτόπου στα Δυτικά Βαλκάνια. Μόνο με συγκεκριμένα αποτελέσματα θα πείσουμε αυτού οι οποίοι αμφιβάλλουν για τον διεθνή ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος του κύριο Βαντάλεν. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η Ολλανδία και τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ένωσης αμήνονται αυτή τη στιγμή στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Και θέλω να το κρατήσω αυτό, να παραμείνει. Σε αυτή τη συνεργασία τα εθνικά κοινοβούλια είναι εκείνα που αποφασίζουν αν θα στείλουν στρατεύματα σε επικίνδυνες περιοχές, άνδρες και γυναίκες των ενόπλων των δυνάμεων. Και η χώρα μου ε, κοντεύει να πιάσει το 2% που ζητάει το ΝΑΤΟ. Δε γιούρε όμως, πουθενά δεν λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ευρωστρατός. Αλλά de facto, στην παράγραφο 116, 118 και 120 γίνεται λόγος για ένα τέτοιο ευρωστρατό. Και μου φαίνεται λίγο περίπλοκο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το ΝΑΤΟ και ευτυχώς ε, ε, γίνεται όλο και πιο σημαντικότερο και θέλω να παραμείνει. Ο κύριος Φουρλάς έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να πάρουμε θέση στο υποσυζήτηση θέμα θα πρέπει να ρωτήσουμε ήδη πρώτα τους εαυτούς μας τι Ευρώπη θέλουμε, τι Ευρώπη χρειαζόμαστε, πώς θέλουμε να φτιάξουμε το κοινό μας σπίτι. Για μένα αγαπητοί συνάδελφοι η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη ισχυρή. Μια Ευρώπη που δεν χρειάζεται τρίτους να εγγυηθούν την ασφάλειά τη διότι μπορεί να το πράξει η ίδια. μια ευρώπη την οποία καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να απειλεί και να εκβιάζει είτε με χτύπημα εναντίον κράτου μέλου είτε με ροέ προσφύγων χωρί επιπτώσει. χρειαζόμαστε μια ευρώπη όπου κάθε κράτο μέλο, όσο μικρό κι αν είναι να έχει ισότιμη φωνή. μια ευρώπη που οι πολίτε θα λαμβάνουν μέρο στι αποφάσει για το κοινό του μέλλον. αυτή την ευρώπη χρειαζόμαστε. για αυτή την ευρώπη πρέπει να αγωνιστούμε αυτή η ευρώπη πρέπει να είναι το κοινό μέλλον όλων μας. ευχαριστώ πάρα πολύ. Να Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρας, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε Μπορέλ, μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις. Και η εικόνα που δόθηκε σήμερα στη συζήτηση για το Ιράκ και το Ιράν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε μια τέτοια συζήτηση για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και πολιτική ασφάλειας, τι εικόνα δίνουμε. Είχατε καθίσει προηγουμένως στη θέση τη Κομισιόν και τώρα αλλάξατε θέση και πήγατε στα έδρανα του Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία. Και αυτή η εικόνα εκφράζει ε, το πόσο διχασμένοι είμαστε. Και όταν είμαστε διχασμένοι δεν είμαστε αξιοπιστοί, ούτε αποτελεσματικοί. Και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλετε να είναι η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίω και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει γεωπολιτική διάσταση, ε, τότε χρειαζόμαστε μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Κάντε ό,τι μπορείτε για να γίνουμε μια αμυντική ένωση, μια ένωση ασφαλείας, μια πολιτική ένωση. Σε αυτή την αντιπαράθεση εσείς πρωταγωνιστείτε τερματίστε τέλους αυτό το πηγαίνω έρχομαι στα διάφορα ε, ε, έδρανα και έχω διάφορους ρόλους και αξιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χριστοφόρου παρακαλώ. Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να εξάρω την προσπάθεια και πραγματικά είναι άξιση χαρητηρίων οι αγαπητοί συνάδελφοι Νταζάν και Μακάλιστερ για την εξαιρετική έκθεση την οποία διεκπαιρέωσαν θεωρώ ότι ισχυρή άμυνα και ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ένωση είναι το τεράστιο έλλειμμα που κουβαλά στους ώμους της η ευρωπαϊκή ένωση είναι το μεγάλο βαρύδιο είναι το μεγάλο στίγμα και άμυνα και ασφάλεια η ευρωπαϊκή ένωση έπρεπε να έχει χθε. ήδη αργοπορήσαμε. η ευρωπαϊκή ένωση για να μπορέσει να προστατεύσει τα σύνορά τη όπω διακηρύττει και να διαφυλάξει όπω είναι υποχρέωση και καθήκον τη την κυριαρχία των χωρών μελών τη οφείλει να διαθέσει χρήματα από τον προπολογισμό και να αρχίσει από τώρα να χτίζει την άμυνα και την ασφαλειά τη. δεν θα μπορούσε καμία τουρκία να φανταστεί να διανοηθεί να εισβάλλει στη συρία στη λιβύη να κατέχει την κύπρο να εισβάλλει στην κυπριακή αγωz να απειλεί χώρε τη ευρωπαϊκή ένωση εάν υπήρχε αυτή η άμυνα και ασφάλεια τη ευρωπαϊκή ένωση. αλλά θεωρώ ότι μέχρι να φτάσουμε στην ενιαία άμυνα και ασφάλεια οφείλουν οι χώρε μέλη τη ευρωπαϊκή ένωση να αντιδράσουν και θα ήταν ένα καλό βήμα κύριε μπορέλ αν υπήρχε μια πρώτη απόφαση από τις χώρες μέλη στα πλαίσια της αλληλεγγύης να αντιδρούν ενωμένου ενάντια σε οποιαδήποτε επιβολή σε χώρα μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης και παραβίαση της κυριαρχίας της και αυτή η αντίδραση να είναι με όλα τα μέσα. Ευχαριστώ. Ε, Μαυρίδης, ε, η Τόμασιτς, Ντάλι και Σδεμιρά είναι τα Catch the Eye. Πέντε συνάδελφοι θα πάρουν το λόγο. Η κυρία Βίρκουνεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για πολύ καιρό έβλεπε, μάλλον για κάποια χρόνια τώρα πρόσφατα βλέπει την Ευρωπαϊκή, την Ευρωπαϊκή Πολιτική ε, να προχωράει αρκετά γρήγορα. Θα πρέπει όμω να επιταχύνουμε και να είμαστε και πιο ενωμένοι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν ζητάμε να ισχύει ο κανόνα τη ομοφωνία. Γι' αυτό το λόγο είμαι υπέρ αυτού προτείνει ο εισηγητή που πρότεινε ο εισηγητή στην Επιτροπή να περάσουμε στην ενισχυμένη πλειοψηφία για όλα τα όσα θέματα είναι δυνατό αυτό. Όταν δηλαδή, ο κύριο δηλαδή όπου δεν χρειάζεται να τροποποιήσουμε τη συνθήκη. Ε, σε, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε θέματα οικονομίας, ε, σε θέματα κοινωνίας των πολιτών. Εκεί μπορούμε να περάσουμε στην ενισχυμένη πλειοψηφία. Θα ήθελα το μήνυμα να περάσει έτσι ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται πιο γρήγορα και για να είμαστε πιο ισχυροί και αξιόπιστοι στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρίδης, παρακαλώ. Yeah, you were asking for the floor κύριε πρόεδρε καταρχήν τα συγχαρητήριά μου στους δύο εισηγητές συναδέλφους. πριν μερικά χρόνια η διαμόρφωση κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας για την ευρωπαϊκή ένωση θα ήταν μια υπερφιλόδοξη θεωρία. σήμερα οι εξελίξεις και οι συνθήκες της παγκοσμιοποίησης το απαιτούν εάν η ευρωπαϊκή ένωση θέλει να διατηρήσει την οικονομική της σταθερότητα την ευρωστία αλλά και να διασφαλίσει το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο συγκεκριμένα χωρίς ενεργειακή ασφάλεια για παράδειγμα είμαστε ευάλωτοι σε απειλές και εκβιασμούς αλλά η ενέργεια προϋποθέτει προστασία και ασφάλεια από στρατιωτικές απειλές και τρομοκρατικές επιθέσεις. για να υπάρξει ειρήνη δεν αρκεί να το θέλουμε εμείς και δυστυχώς όσοι ακόμα ονομάζουν τον ερντογάν στρατηγικό εταίρο δυστυχώς θα το μετανιώσουν. κύριε Μπορέρ, i'm going say this in english libya syria η Συρία, η Λιβύη, τα κατεχόμενα στη Βόρεια Κύπρο, ε, η Ανατολική Μεσόγειος, ε, όλα αυτά έχουν το ίδιο όνομα. Τουρκία, επεκτατισμός. Κυρία Τόμασιτς. Η έκθεση για την ε, εφαρμογή τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα ε, περιλαμβάνει και την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Ε, τονίζεται ότι αυτό το τμήμα τη Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό για την σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, υπογραμμίζεται ότι μια ισχυρότερη δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται σε αυτό το κομμάτι τη Ευρώπη πέραν των δράσεων του ΟΗΕ. Ναι, είναι προτεραιότητα και για την Κροατία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Πιστεύω όμω ότι σημαντική πρόοδο στα Δυτικά Βαλκάνια δεν θα να, μπορέσει να επιτευχθεί και δεν θα επιτευχθεί μέσω αυταρχικών ε, ηγετών όπως αυτός της Σερβίας ή αγνοώντας ε, τις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κροατικού λαού που συμβαίνουν στην Βοσνία Ρεζεγοβίνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει αλλιώς να συνεισφέρει στη βελτίωση της κατάστασης ε, για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα, να τα κοιτάξουμε στα μάτια και να εργαστούμε γι' αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν είμαι υπέρ της ε, ΚΕΠΑ. Ε, νομίζω ότι αναγκαστήκαμε δύο φορές να ψηφίσουμε γι' αυτό στην Ιρλανδία και πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ πάρα πολύ για τις εξελίξεις στην ΚΕΠΑ και στην ΚΠΑ που έχουν τεράστιες και δυσάρεστες εξελίξεις. Γι' αυτό εμείς θα αντισταθμούμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια να δεχθούμε την ειδική η στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο δεν είναι προς όφελος των πολιτών. Ε, η νέα, μια νέα λευκή βίβλος, αυτό που ζητάει η έκθεση, αυτό θα ήταν ένα νέο βήμα, όχι θετικό βήμα, ένα ε, κάτι το οποίο ζητούν η Γαλλία, 13 ε, καινούργια προγράμματα της μόνιμης διαρθρωτημένης συνεργασίας είναι γαλλικής έμπνευσης έτσι ώστε να στρατιωτικοποιηθεί η Ευρώπη Ευρώπη, αγνώντας βέβαια το τι συμβαίνει με τη συντάξη στη Γαλλία. Γι' αυτό δεν πρέπει να επεμβαίνουμε σε άλλες χώρες. Πρέπει να αναφέρετε το άρθρο 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπου προβλέπεται το να διαφυλάσσονται ε, τα ε, κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, αυτά ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Κυρία Πρόεδρε, η ΠΕΣΚΟ, η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, τα στρατεύματα και το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο, αυτά είναι ε, συνθήματα, λέξεις κλειδί και νομίζω είναι απόλυτα σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να περικόψει τα κοινωνικά προγράμματα και να δώσει πάρα πολλά χρήματα, δισεκατομμύρια στα λόμπι. Κυρίε και κύριοι, ε, παραβιάζεται το ενωσιακό δίκαιο. Το 1-2 ε, λέει ότι οι δαπάνε από την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να δίδονται για στρατιωτικά μέσα. Είναι αλήθεια ότι ο, η κατάσταση είναι πολύ ευαίσθητη, πάρα πολλέ συγκρούσει. Απλά όμω να τα αναφέρει κανεί αυτά στην έκθεση χωρί να εξηγεί και τον ρόλο των κρατών μελών, αυτό είναι υποκρισία. Η εμπορική πολιτική, οι εξαγωγέ όπλων από τα κράτη-μέλη σε αιστείε κρίση, αυτά όλα οξύνουν τι συγκρούσει. Αν σα ενδιαφέρει η ειρήνη και η δημοκρατία, θα πρέπει να στείλετε το, τις εξαγωγές όπλων σε ολόκληρο τον κόσμο, να μην υπάρχει αυτό το σπιράλ των εξοπλισμών, δεν θα πρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να τη μετατρέψετε ε, σε μια στρατιωτική ένωση. Να περιορίσετε τους εξοπλισμούς, αυτό θεωρώ ότι είναι μια βιώσιμη πολιτική ασφάλειας και όχι αυτό που κάνετε εσείς, γιατί αυτό που κάνετε εσείς είναι πραγματικά θανάσιμα επικίνδυνο. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ε, Αντιπρόεδρο, τον ε, κύριο ε, Μπορέλ. Έδινα κάποιες οδηγίες γιατί έξω από την αίθουσα ο κόσμος εξακολουθεί να γυρίζει και συμβαίνουν διάφορα. Πρέπει να ευχαριστήσω τους δύο, τους δύο συγητές Πιστεύω ότι και οι δύο είναι πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις. Ε, ανοίγουν μια, μια σημαντική συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιος είπα ότι άλλαξα από τα έδρανα της Κομισιόν πέρα στα έδρανα του Συμβουλίου. Ναι, ναι. Εκείνη η Κομισιόν και εδώ είναι το Συμβούλιο, πράγματι. Και γνωρίζετε ότι ο ύπατος εκπρόσωπος εκπροσωπεί και το Συμβούλιο, εκπροσωπεί το Συμβούλιο αλλά με έδρα την Κομισιόν. Και όσο είναι έτσι τα πράγματα θα πρέπει να αλλάξω, να αλλάζω θέση. Αν θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση πρέπει να αλλάξουμε τη συνθήκη. Και σίγουρα δεν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα. Θα χρειαστούμε λίγο περισσότερο χρόνο. Δεν καταλαβαίνω τους φόβους κάποιων κρατών ότι θα δημιουργήσουμε ένα τέρας ε, στρατιωτικό τέρας και θα πέσουμε σε, κάποια, ε, σε κάποιους φεντεραλιστικούς γκρεμούς. Δεν καταλαβαίνω. Η Κομισιόν που είναι ένα όργανο που βοηθάει στην ομοσπονδοποίηση, α το πούμε έτσι, δεν έχει αρμοδιότητε σε θέματα Άμυνα και ασφάλεια. Οπότε θα ρωτήσει κανεί γιατί δημιουργούμε την αμυντική ένωση εφόσον δεν έχουμε αρμοδιότητες. Ε, η αμυντική ένωση έχει σχέση με την, ε, όχι με την ίδια την άμενα, αλλά με την αμυντική βιομηχανία. Γι' αυτό, είτε το θέλουμε είτε όχι, ζούμε σε έναν κόσμο που η κοινή εξωτερική πολιτική την χάνει διαχείριση από το Συμβούλιο με ομοφωνία. Πολύ μακριά από την ομοσπονδοποίηση. Τι τύπου ομοσπονδία είναι αυτή το ίδιο σημαίνει και με την πολιτική άμυνας. Οπότε δεν καταλαβαίνω τους φόβους κάποιων ότι θα πέσουμε στη μαύρη τρύπα του φεντεραλισμού. Είμαστε παρασάγκας απέχουμε από αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη να εμβαθύνει την διάσταση της ε, κοινή δράσης στον κόσμο. Το πιστεύω ειλικρινά. Υπάρχουν κάποιοι εδώ, μέλη του Κοινοβουλίου, που δεν το πιστεύουν. Εγώ προσωπικά το πιστεύω και όταν ήμουν υποψήφιος ε, να γίνω επίτροπος, το υποστήριξα στις ακρόασεις. Θα πρέπει να είμαστε ικανοί να δρούμε με πιο αποτελεσματικό και ισχυρό τρόπο σε ένα πολύπλοκο κόσμο, σε μια πολύπλοκη διεθνή σκηνή. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ε, ακολουθούμε <clears throat> κοινή στάση. Κοινή στάση δεν σημαίνει <clears throat> μοναδική στάση. Δηλαδή είχαμε ένα κοινό νόμισμα που δεν ήταν το μοναδικό. Δηλαδή είχαμε ένα κοινό νόμισμα και κάποιοι είχαν το δικό τους νόμισμα. Για κάποια πράγματα δουλεύουμε όλοι μαζί και για κάποια άλλα ο καθένας μόνος του. Πόσο χρόνο χρειαστήκαμε για να περάσουμε από το κοινό νόμισμα στο ενιαίο μοναδικό νόμισμα. 20 χρόνια, Μ, ίσως παραπάνω. Το νόμισμα που είναι σύμβολο εθνικής κυριαρχίας δεν είναι το πιο ισχυρό. Η άμυνα, η ειρήνη, ο πόλεμος η ικανότητα να προασπίζουμε τα συμφέροντά μας στον κόσμο είναι πολύ πιο κοντά στην κυριαρχία. Οπότε θα χρειαστούμε ακόμα περισσότερο χρόνο για να περάσουμε από την κοινή πολιτική στην ενιαία πολιτική. Και αυτή η έκθεση δείχνει πολύ καλά ποιε είναι οι δυσκολίε. Και εγώ το ζω σε πρώτο πρόσωπο. Όταν συζητάμε για μια χώρα που είναι τόσο κοντά σε εμά, τη Λιβύη, βλέπουμε πόσο διαφορετικές είναι οι εθνικές θέσεις. Και αυτή είναι η αδυναμία μας. Οπότε ο δρόμος θα είναι μακρύ. Αλλά θα πρέπει να αποκτήσουμε κοινέ στρατιωτικές ικανότητες έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε όχι με ομοφωνία αλλά με ε, ενισχυμένη πλειοψηφία. Και αυτή η έκθεση δείχνει το δρόμο κατά κάποιο τρόπο και τις δυσκολίες. Γι' αυτό το λόγο χαιρετίζω, χαιρετίζω και τις δύο εκθέσεις. Ευχαριστώ τους συζητητές και ελπίζω ότι θα συζητήσουμε ακόμη περισσότερο από κοντά ε, γιατί μόνο έτσι θα ενισχύσουμε τη θέση μας στον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να λύσουμε όλα τα προβλήματα του κόσμου όντας εντός των συνόρων μας όλα τα προβλήματα χρειάζονται διαβήματα εκτός των συνόρων μας. Η μετανάσταση, η μετανάστευση, η πόλεμη, όλα είναι γεωπολιτικά σήμερα, είναι η λέξη της μόδας. Και για να είναι κανείς γεωπολιτικός παίκτη, θα πρέπει να έχει στρατιωτικές ικανότητες και διπλωματικές ικανότητες και συχνά λέμε ότι θα πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ του να είμαστε παίκτη, player ή να είμαστε γήπεδο. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να... ότι είμαστε ήδη παίκτη, αλλά αναζητούμε ακόμα την ταυτότητά μας. Δεν ξέρουμε τι είδου παίκτη είμαστε. Με εκθέσεις σαν κι αυτές μπορούμε να εμβαθύνουμε σε αυτό το υπαρξιακό ερώτημα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ ε, όλα τα μέλη για τη συμμετοχή τους. Κρίμα που δεν έχουμε μεγάλα πλήθη να ενδιαφέρονται για μια συζήτηση τέτοιας ύψης της σημασίας. Αλλά πάντως ευχαριστώ πολύ που μείνατε εδώ μέχρι τόσο αργά και παρακολουθήσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα και κρίσιμη για το μέλλον μας συζήτηση, για το μέλλον μας ως κοινωνία σε έναν ταραχώδη κόσμο. Ευχαριστώ πολύ κύριε είπατε εκπρόσωπε και τώρα θέλω να σας ευχαριστήσω ε, για τους επένους και εξ ονόματος των δύο εισηγητών, στους οποίους θα δώσω και το λόγο. Κύριος Μακάλιστερ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, ο υπατός εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος μόλις μίλησε για πολλά θέματα και επειδή έχει περάσει και η ώρα, θα πρότεινα να μείνω σε πολύ λίγα. Θα είμαι πολύ σύντομος να σας ευχαριστήσω όλους για τις συνεισφορά για την ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση που είχαμε. Χάρηκα που άκουσα την πλειονότητα των ομιλητών να συμφωνεί με ε, την πρότασή μας για μια πιο ισχυρή κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ακόμα έχουμε στο μυαλό μας τις συζητήσεις που επίκενται για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και κύριε Μπορέλ θα πρέπει να εξασφαλίσετε όχι απλώς ε, τη χρηματοδότηση αλλά τη συνέπεια, τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα και την ευθύνη των μέσων αυτών για την εξωτερική πολιτική. Θέλω να σας ευχαριστήσω. που παρέμεινε όλες αυτές τις ώρες εδώ στο ημικύκλιο και δείχνει το σεβασμό του προς το Κοινοβούλιο. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς παρόντε εδώ, τόση ώρα είναι και ο ίδιος. Ο κύριος Ντανζάν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή. Πολλές ενδιαφέρουσες ομιλίες ακούσαμε. Λυπάμαι που ορισμένοι προχωρούν σε δίκη προθέσεων. Οι εκθέσεις μας δεν είναι ιδεολογικά φορτισμένες. Είναι αρκετά ρεαλιστικές εκθέσεις. Κατα... Αναδεικνύουν μία πραγματικότητα. Ζούμε σε πολύ ταραγμένο κόσμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει το ρόλο της εκεί και το στρατιωτικό της ρόλο. Ακούω συναδέλφου που αγανακτούν για τη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μύθος είναι αυτό, εφιολόγημα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θα πρέπει να εξορροπήσουμε στην πολιτική ασφάλεια και ε, ε, ανάμεσα στο στρατιωτικό και το πολιτικό σκέλος. Αν το κάνουμε αυτό και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή του στρατιωτικού σκέλους. Γιατί σήμερα ουσιαστικά η συνεργασία μόνο πολιτική είναι. Έχουμε 11 αποστολέ πολιτικής φύσεως και 5 στρατιωτικής φύσεως. Προσοχή για αυτά που λέμε. Η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς αυτή που κάποιοι συνάδελφοι περιγράφουν. Και είναι λίγο κρίμα αυτό. Γιατί εγώ ε, είχα κάποιες ευθύνε. Ε, σε κάποιες ε, ζώνες κρίσεων που είναι παρούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα κάποια ταπεινή συμμετοχή κι εγώ ε, και πήγα και έμαθα τι γίνεται, τι κάνει η Κομισιόν, τι κάνουν τα κοινά στρατεύματα, οι αποστολές, οι εθνικές αποστολές. Χρειάζεται η Ευρώπη, ας είμαστε ρεαλιστές και στους συναδέλφους που, που ανησυχούν μήπως απαγκιστρωθούμε από το ΝΑΤΟ. Μα δεν πρόκειται κανείς να αντικαταστήσει το ΝΑΤΟ για τη συλλογική ασφάλεια, αλλά υπάρχουν μέρη που δεν έχει συμφέρον το ΝΑΤΟ να επέμβει. Άκουσα στην αρχή της εβδομάδας τον πρόεδρο Τραμπ να ανακοινώνει ότι ε, θα ε, αποσυρθούν δραστικά από την Αφρική, από τη Σομαλία, τον Ήγηρα και το Μάλι τα αμερικανικά στρατεύματα. Τι θα κάνουμε. Εμείς ε, θα υπολογίζουμε στους Αμερικανούς, μα θα πρέπει να μπορούμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Το είπα και εισαγωγικά. Υπάρχουν κάποια μέρη του κόσμου που δεν έχουμε τις ίδιες προτεραιότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε ε, ε, σύμμαχοι. Ούτε αναθεωρούμε, ούτε αμφισβητούμε την παραδοσιακή μας σχέση. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι υποτρεδιότητές μας και τα συμφέροντά μας εκεί που κάποιοι άλλοι αποχωρούν. Αν δεν θέλουμε να χαθούμε από το γεωπολιτικό χάρτη, θα πρέπει να αναλάβουν με αυτή μας την ευθύνη. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Πριν προχωρήσουμε με το επόμενο θέμα που είναι η κατάσταση στη Λιβύη, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λήφθηκαν κάποιες αποφάσεις για ορισμούς σε πολιτικές ομάδες και σε ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αυτά αναφέρονται στα σημερινά ε, συνοπτικά πρακτικά και τίθεται σε ισχύ από σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και ε, για το έργο σας. Αυτό προς τους εισηγητές τους δύο. Θα κάνουμε πέντε λεπτά διάλειμμα για να μπορέσουν λίγο να ξεκουραστούν όλοι οι συμμετέχοντες στη συζήτηση. Συνεχίζουμε σε πέντε λεπτά.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 λόγο για την μπλε κάρτα, τη νέα ηλεκτρονική. Ουσιαστικά ένα κουμπί πατάτε, είναι πάρα πολύ απλό. Θα δώσω το λόγο για πέντε λεπτά τώρα, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπορέλ. Ακολουθεί ο κύριος Μακάλιστε και μετά η κυρία Πύρη. Εξ ονόματος των πολιτικών του ομάδων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα πράγματα στη Λιβύη πάνε από το κακό στο χειρότερο. Ίσως τις επόμενες μέρες να δούμε κάποια ακτίδα φωτός, ελπίδας, αλλά από τα Χριστούγεννα οι επιθέσεις ε, των, του στρατού του Χαφτάρ ε, εντάθηκαν βομβαρδισμοί εναντίον αμάχων το ίδιο ε, δολοφονία 30 μαθητών της ε, Στρατιωτικής Ακαδημίας στην Τρίπολη μια επίθεση την οποία καταδικάσαμε αλλά δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να καταδικάζουμε επιθέσεις ο πόλεμος αυτός είναι πόλεμος κατεξιοδότηση και έχει ένα αριθμό θυμάτων πραγματικά είναι απαράδεκτος. Και 350.000 ε, άτομα άμαχοι που έχουν μετακινηθεί, ε, έχουν εγκαταλείψει αιστείες τους κοντά στην Τρίπολη. 300 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους, χιλιάδες ε, θύματα στρατιωτικοί, επιθέσεις σε